Έχουμε αρκετά μέλη παρόντα και μπορούμε να αρχίσουμε καταρχάς με την έγκριση της μερίσιας διάταξης. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Είναι κρίμα που οι ανακοινώσει για τον τριμερή διάλογο γίνονται πάντοτε με κενά καθίσματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υποθέτω μας, ακούμε, μας ακούν από το διαδίκτυο. Λοιπόν, ανακοινώσει της Προέδρου 2013-2017 ε, στατιστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανόνα, κανονισμό 73 και σας ενημερώνω η τελική διαδικασία, τα τελικά τμήματα έγινε με γραπτή διαδικασία και έχουμε συμβαστική πρόταση του Συμβουλίου και αν δεν υπάρχει αντίρρηση από τις ομάδες κατά τη διάρκεια αυτής της Επιτροπής, μια ένα συμβιβαστικό σχέδιο έκθεση θα υποβληθεί στον Ολομέλεια του Ιανουαρίου και ήθελα να ευχαριστήσω τον Έντουαρτ Σεκλούνα για τη διεξαγωγή όλης αυτής της διαδικασίας για την ε, οδηγία κεφαλουχικών ε, υποθέσεων κριτηρίων ε, θα συζητήσουμε τα θέματα της ρευστότητα, τα ομόλαγα και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών και τη διαχείριση κρίσεων. Έχουμε ταυτοποιήσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ε, προτάσεις στην ε, τεχνική ομάδα εργασίας. Ο επόμενος ε, το ημερής διάλογος θα γίνει στις 12 ενδεκάτου και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Κατά την πράσινη εβδομάδα, μία αντιπροσωπεία της ΣΥΚΟΝ πήγε στην Ιταλία από την προεδρία του Αντιπροέδρου Πιερτό Στόγιαν και οι συζητήσεις που έγιναν εκεί ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικέ με εκπροσώπους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των ε, ρυθμιστικών αρχών. Ε, συζήτησαν για τα θέματα της Ιταλικής οικονομίας και έχουν μία, ένα ανακοινωθέν τύπου, τύπου και σας παραπέμπω σε αυτό για περαιτέρω λεπτομέρειες. Επίσης, σας προτείνω, σας συστήνω ε, σας ενημερώνω ότι ο Πρόεδρος επανέλαβε την ε, πρόσκληση αυτή για έναν ε, διάλογο τριμερή με τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικών που μπορεί να γίνει πριν το τέλος του χρόνου. Έτσι ολοκλήρωσα τις ανακοινώσεις της Προέδρου και τώρα θα ήθελα να αρχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Hans Hogervorst, πρόεδρο του Συμβουλίου Δεχνολογιστικών Λογιστικών Είναι η πρώτη του επίσκεψη εδώ και όπως ξέρετε έχει μία μακρά εμπειρία στα λογιστικά πρότυπα ε, και ε, εμπειρία επίσης για όλα στις πτυχές της τραπεζικής σταθερότητος, των προβλημάτων κλπ. Και θα ήθελα να μας παρουσιάσετε, να μας κάνετε την εισαγωγή σας και μετά θα έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις.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 στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου σήμερα, θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένες από τις παρατηρήσεις και τις ε, ερωτήσεις σας. Ενδεχομένως να έχει έρθει σε επαφή Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της μίσθωσης που πάρα πολλές φορές ομοιάζει με δάνειο και πολλές φορές δεν εμφανίζεται με τον σωστό τρόπο στον ισολογισμό των εταιριών. Η συνολική παγκόσμια αγορά μίσθωσης αντιστοιχεί σε 600 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία παραμένουν εκτός ισολογισμού τις περισσότερες φορές. Εμείς θέλουμε οι επενδυτές να είναι σε θέση να δουν ότι υπάρχει αυτή η πραγματική αλλά κρυμμένη μόχλευση. Και εφόσον η χρηματοπιστωτική κρίση δημιουργήθηκε από ένα υπερβολικό χρέος, θα θέλαμε και τη δική σας τη βοήθεια προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να αποδίδουμε καλύτερα στους ολογισμούς το ζήτημα της μίσθωσης. Η δεύτερη πρόκληση που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε έχει να κάνει με το τι θα κάνουν τελικά οι Ηνωμένε Πολιτείε με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαίου των Ηνωμένων Πολιτείων υποστηρίζει την εργασία μας τελευταία χρόνια. Το 2007 η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαίου αναγνώρισε την υψηλή ποιότητα των διεθνών λογιστικών προτύπων και επέτρεψε σε ε, διάφορες εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο Αμερικανικό χρηματιστήριο να χρησιμοποιούν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αμερικανική αγορά. Has not been made yet. The SEC had intended to make this decision in 2011, but announced in July that it would postpone this decision yet again. That was really disappointing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 and which will force banks to recognize unavoidable losses at a much earlier stage than is currently the case. This is, I think, the most important. Πιστεύω ότι είναι η πιο μεγάλη αλλαγή στους κανόνες λογιστικής η οποία λαμβάνει η χώρα. Και είναι ο, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Υπάρχει κάποιος από τη σοσιαλιστική ομάδα που θα ήθελε να λάβει το λόγο, Αντολίν. Ευχαριστώ πολύ. Σε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και πιστεύω ότι η σύγκληση στα θέματα των λογιστικών προτύπων είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα ώστε να μπορέσει να γίνει απαραίτητη μεταρρύθμιση στα θέματα κανονιστικής ρύθμισης. Για όλα αυτά τα ζητήματα η διαδικασία αυτή έπρεπε να έχει τελειώσει τον ε, Ιούνιο του 2011, αλλά στις ε, συζητήσεις των G20 υπάρχουν συνεχεία μνήες στην ανάγκη να συνεχιστούν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα θέματα τα οποία παραμένουν εκκρεμή, αν είναι εκκρεμή μέσα σε μια ημερήσια διάταξη ή αν είναι εκκρεμή στο, διηνεκή, στο τα θέματα αυτά. Ποια είναι ακριβώς τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Επίσης θα ήθελα να ξέρω αν υπάρξει αυτή η σύγκληση θα πρέπει ο φορέας ο οποίος θεσπίζει τα πρότυπα αυτά να είναι και αυτός αντικείμενο κάποιας ε, σύγκλησης. Θα ήθελα λοιπόν αν έχετε κάποια να μας πείτε σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του πολυμερούς φορέα στο μέλλον και ποια ακριβώς είναι η σύνθεσή του. Μία ακόμα ερώτηση. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαφάνεια, ιδίως η διαφάνεια σε σχέση με εξορρυκτικές δραστηριότητες δραστηριότητε οι οποίε αφορούν την εκμετάλλευση φυσικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο μα. Λένε πολλέ φορέ και να προχωρήσουμε περισσότερο στον τομέα αυτό θα είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια προσέγγιση, μια μεγαλύτερη σύγκληση σε σχέση με τα λογιστικά πρότυπα. Τι προβλέπετε να γίνει στον τομέα αυτό. Thank uh, Σας ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα που μου θέσατε. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε, ότι η σύγκληση δεν έχει επιτευχθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που είχαμε ελπίσει. Αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία όταν υπάρχουν δύο τέτοιοι φορείς, ένας παγκόσμιος φορέας και ένας αμερικάνικος τομέας, αμερικάνικος φορέας. Φανταστείτε την Βασιλεία τρία να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση από δύο χωριστέ επιτροπές Δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει. Η ύπαρξη λοιπόν δύο φορέων για τα λογιστικά πρότυπα οδηγούν, οδηγεί σε προβλήματα σε σχέση με την υλοποίησή τους. Επίσης, οι ΗΠΑ δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε μία απόφαση για να εγκρίνουν το IFRS. Τα διεθνή πρότυπα χρηματοπιστωτικής αναφοράς. Και εξακολουθεί να γίνεται δύσκολο και να είναι δύσκολο να συμφωνήσουν οι Αμερικανικοί φορείς μαζί μας. Έχουμε δει στην περίπτωση που ανέφερα προηγουμένως το μοντέλο της προσδοκόμενης απώλειας. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα στα οποία είχαμε καταφέρει να επιτύχουμε κάποια σύγκληση και τον Ιούλιο του 2012 υπήρξε από την Αμερικανική πλευρά μια διαφωνία. Είπαν ότι δεν θα ακολουθήσουν το δικό μας μοντέλο, αυτό το μοντέλο που ήταν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων και θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Ε, επομένως δεν είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ακολουθήσουν το ίδιο δρόμο μαζί μας στο άμεσο μέλλον. αυτά στα οποία έχουμε επιτύχει κάποια σύγκληση είναι το θέμα της μίσθωσης και της αναγνώρισης των ε, εσόδων. Εκεί υπάρχει κάποια προσέγγιση για τις ε, συμβουλευτικές ομάδες πολυμερούς χαρακτήρα. θέλαμε καταρχήν να εξασφαλίσουμε μια μείωση των, ε, της σύνθεσης αυτών των φορέων σε 12 άτομα. Θέλουμε να έχουμε πραγματικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα αποδίδονται σε συζητήσεις σε βάθος. Επομένως δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο αυτό το σώμα σε σύνθεση. 12 είναι ένας φυσικός αριθμός. Τώρα ποιοι θα είναι μέλη αυτού του φορέα δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Αλλά έχουμε τώρα περιφερειακές ενότητες στον κόσμο. Έχουμε μια περιφερειακή ομάδα που περιλαμβάνει την Ασία και την ε, Αμερική και, Νότια, και Νέα Ζηλανδία. Έχουμε τον φορέα τον Ευρωπαϊκό. Έχουμε μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής που αφορούν τα θέματα προτύπων. Όλοι αυτοί οι φορείς που σε περιφερειακό επίπεδο εκπροσωπούν μια πλειάδα χωρών θα είναι αυτόματα μέλη. Στη συνέχεια θα προσκαλέσουμε ε, μεμονωμένους εκπροσώπους, χάρη από την Ιαπωνία, Ίσως από κάποια ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος εκπρόσωπος και θα υπάρξει και εκπεριτροπής κατάληψης των θέσεων σε αυτό το φορέα, ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν καιρό. Αυτή τη στιγμή όμως απλώς προσπαθούμε να καταρτήσουμε τις αδρές γραμμές για αυτόν τον φορέα. Και όλα εξαρτώνται από τις ανταλλαγές απόψεων που θα έχουμε με τους φορείς μας ο καθένας. Για το θέμα τώρα της διαφάνειας, νομίζω ότι αναφέρεστε στις, ε, στις εκθέσεις που αφορούν κάθε χώρα μεμονωμένα. Σας είχα πει ότι θα κοιτάξουμε την ανάγκη να υπάρξει μια νέα διαβούλευση, εάν υπάρχει πρόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, για να είμαι ειλικρινής δεν υπήρξε πάρα πολύ θέληση σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των μελών μας για μια νέα διαβούλευση για τα θέματα αυτά και από ό,τι κατανοώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μέσα σε ένα αριθμιστικό πλαίσιο να προχωρήσει τα πράγματα και ίσως αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να επιτύχουμε κάποια πρόοδο. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να επιτύχουμε πλήρως το στόχο αυτό. Βλέπω στις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν τα θέματα αυτά μετά το νόμο Dodd-Frank και η Ηνωμένη Ευρώπη επίσης προχωρεί προς την κατεύθυνση αυτή και υπάρχει έτσι κάποια ελπίδα. Ο Βόλφ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ που έρχεστε εδώ για δεύτερη φορά και που έχετε δηλώσει την προθυμία σας ε, εδραίωσης ενός τακτικού διαλόγου. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει πάση θυσία να επιδιώξουμε τη σύγκληση εάν δεν, μπορούμε να, εάν δεν γίνεται να επιτευχθεί επειδή υπάρχουν αντι, αντίθετα κριτήρια και προδιαγραφές, εντάξει, έστω. Όμως πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε στρεβλώσεις. Παραδείγματος χάρη, εισαγωγή της Βασιλείας 3, παρόλο που υποτίθεται την υποστηρίζουν οι Αμερικανοί, ε, έχει δημιουργήσει ορισμένες ετήσιες ε, δαπάνες, όμως στην Αμερική τα ίδια κονδύλια τα οποία για μας θεωρούνται ως δαπάνες, στην Αμερική αποσβαίνονται. Αυτό δημιουργεί έναν ε, στρεβλό ανταγωνισμό, μια στρέβλωση της κατάστασης και το ερώτημά μου είναι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να, να ξεπεράσουμε αυτή την ακραία περίπτωση, το ακραίο παράδειγμα. Διαπιστώνουμε επίσης ότι σήμερα έχουμε ένα σωρό οικονομικά, χρηματοοικονομικά κέντρα, τα οποία θα αυξάνουν την ισχύ τους τα επόμενα 20-25 χρόνια. Μουμπάι, Σανγκάι, Χονγκ Ντουμπάι, μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Είναι λοιπόν σημαντικό εκεί όπου προσπαθούμε να εδραιώσουμε διεθνή πρότυπα να μπορέσουμε και να τα εφαρμόσουμε, να είναι εφαρμόσιμα. Πολλές φορές κάνουμε συζητήσεις με κοινού στόχους, όμως την υλοποίηση διαπιστώνουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας, μεγάλη απόσταση τι μπορούμε να κάνουμε στα, σε, αυτά τα, σε αυτές τις ομάδες που επεξεργάζονται αυτά τα προβλήματα του G20, IOSCO, FSB, πώς μπορούμε να επιτύχουμε εκεί μια συμφωνία, μια ε, συνένεση. Ευχαριστώ κύριε Κλίντς για αυτές τις ερωτήσεις σας. Δύο σημαντικά θέματα σήξατε. Θεμητό ανταγωνισμό, σε θεμητό επίπεδο παιχνιδιού και ε, συνένεση. Όσον αφορά το δίκαιο και θεμητό, δίκαιη και θεμητή ε, δραστηριότητα, ε, νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος όλων μας. Δύο, σε δύο θέματα έχω πραγματικά απογοητευτεί που δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε σύγκληση. Το ένα ήταν... The e at that Εμπόδια οι αδυναμίες που παρουσιάστηκαν και το δεύτερο είναι ότι όλα τα παράγωγα, ζητήσαμε από τις τράπεζες να παρουσιάζουν όλα τα παράγωγα στον ισολογισμό. Εκεί σε αυτά τα δύο θέματα δεν μπορούσαμε καθόλου να επιτύχουμε σύγκληση. Πιστεύουμε ότι αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία Warren Buffett έχει χαρακτηρίσει ως όπλα μαζικής καταστροφής ε, θα παρουσιάσουν κάποια λύση. Είχαμε λοιπόν προτείνει ακριβώς να παρουσιάζονται τα παράγωγα αυτά τα derivatives στους ισολογισμούς των τραπεζών όμως τελευταία, στην τελευταία στιγμή αυτό δεν εγκρίθηκε. Πιστεύω ότι η λύση που πρότεινε το IFRS δεν συγκρίνεται με τη δική μας. Ε, διότι η άποψη η δική μας λέει ότι ποτέ δεν μπορεί κανείς να είναι αρκετά διαφανής. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να τα δείχνουμε να εμφανίζονται τα πάντα. Προσπαθούμε λοιπόν να εναρμονίσουμε ε, την ε, διαφάνεια, την δημοσιότητα, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να μπορεί να δει παραδείγματο χάρη τι το συμφέρει, η Deutsche Bank ή η JP Morgan, να υπάρξει ένα, σεμιτό, ένα διαφανές και ισοδύναμο πεδίο ανταγωνισμού. Εν συνεχεία, η υιοθέτηση παγκοσμίω. Ε, χαίρομαι που αναφέρεται ορισμένα τεράστια οικονομικά κέντρα, το Σαν Πάολο παραδείγματος χάρη στη Βραζιλία επίσης. Ε, τα, περισσότερα έχουν ήδη πλήρως αποδεχθεί τους, ε, καταπρότυπα πρότυπα του IFRS. Η Σιγκαπούρη, επίσης, πολύ σημαντικό οικονομικό κέντρο, χρηματοοικονομικό κέντρο, όχι, δεν έχει υιοθετήσει απολύτως όλα τα πρότυπα, αλλά σύντομα θα το κάνει άλλες χώρες που ανέρχονται ε, η Δονησία α πούμε, εντάξει, μπορεί να μην γίνει ένα τεράστιο χρηματοοικονομικό κέντρο, αλλά και αυτοί θα υιοθετήσουν. Η Κίνα θα γίνει, θα γίνει και αυτή με τον καιρό ένα μεγάλο, σημαντικό οικονομικό κέντρο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σε εμά αυτέ οι χώρε του IFRS. Αλλά βέβαια θέλουμε να πάρουμε και τις Ηνωμένε Πολιτείε μαζί μας, το πλευρό μας. Είναι μια απόφαση όμως που μόνο οι Αμερικανοί μπορούν να πάρουν για τον εαυτό τους και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε επιρροή. Ένα είναι σαφές ότι οι Αμερικανοί το δέχονται αυτό, ότι ε, ο μόνο υποψήφιο που μπορεί να εδραιώσει πραγματικά διεθνή πρότυπα είναι το IFRS. Και είμαι πεπισμένος ότι είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον των ΗΠΑ να έρθουν και αυτοί, να ανέβουν και αυτοί στο τρένο, το δικό μας. Είναι μια δύσκολη εποχή οικονομικά για όλους. Είναι δύσκολο να πείσουμε εταιρείε να αλλάξουν τα συστήματά τους. Σαφώς θα υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά στο τέρος θα μπορέσουν και οι Αμερικανοί να έρθουν στο πλευρό μας. θα υιοθετήσουν και αυτοί. Η πρόεδρος. Εντάξει. Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Καμάλ, και ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Βεβαίως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διαφάνεια. Ε, ο συνάδελφος μου ζήτησε, ε, ρώτησε πριν τι γίνει με τι, θα, τι γίνεται με τις εκτιμήσεις οι οποίες είναι υπερβολικές είτε είναι υποτιμημένες. Παραδείγματο χάρη η RBC, Royal Bank of Scotland, η οποία είχε εκτιμηθεί σε 25 δις, ε, απεδείχθη ότι είχε υπερεκτιμηθεί και έγιναν και ανάλογες δηλώσεις στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πραγματικά μεγάλες προκλήσεις να υιοθετηθούν ε, το, τα, τα, λογιστικά πρότυπα μέσω του IFRS ως ε, τα ως οι θεμελιώδεις αρχές της λογιστικής. Όμως μπορεί αν εξετάσουμε σε βάθος ε, τους κανονισμούς και τα πρότυπα το IFRS να μην είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, πιστεύετε ότι δικαιολογείται η δυσπιστία προς το IFRS ενδεχομένως δηλαδή να μην αντιπροσωπεύει τα πιο δίκαια λογιστικά πρότυπα. Πο, πολλές φορές υπάρχει υπερβολική ε, η προθυμία υιοθέτηση προτύπων έτσι ώστε να μπορούν να προβλεφθούν όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα επίγοντα και τα ξαφνικά γεγονότα που συμβαίνουν. Γιατί να μην έχουμε ένα περιθώριο ευελιξίας. Παραδείγματο χάρη η AIG ε, κατάφερε να έχει ε, χρέη 3,1 δισεκατομμύρια ε, με τα dealings που έκανε στα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις και να μην είναι όλα τσιμεντωμένα. Σας ευχαριστώ για αυτά τα κέρια ερωτήματά σας. Και εγώ έχω σκεφτεί για τα ζητήματα αυτά αρκετά. Προηγουμένως, σας είπα, υπομορφή σχολείου ότι αν οι ρυθμιστές και οι επενδυτές είχαν προσέξει τα αριθμητικά στοιχεία ήταν πραγματικά φανερό, κατάδειλο ότι οι τράπεζες είχαν πολλά προβλήματα. Η Royal Bank of Scotland είναι ένα από τα πιο χτυπητά παραδείγματα και η ING στην δική μου χώρα. Εγώ ήμουν τότε ε, ρυθμιστής για τα θέματα των αξιογράφων στι κατοχώρε. και δεν κατάλαβα, δεν μπόρεσα να καταλάβω πώ ήταν δυνατόν να υπάρξει μια τέτοια κατάρρευση. Επομένω, νομίζω ότι το πιο απλό θα ήταν να κοιτάξει κανεί του αριθμού και κοίταξα όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Και είδαμε ότι η Royal Bank of Scotland ουσιαστικά δεν είχε ε, κεφάλαιο, είχε μόκλευση 14-15 φορέ. Το κεφάλαιό του ήταν ουσιαστικά αέρα ήταν ε, φήμη και πελατεία ουσιαστικά από προηγούμενες εξαγορές τραπεζών. Κάθε φορά υπερεκτιμούσαν την, ε, την αξία της, ε, της τράπεζας και ουσιαστικά το κεφάλαιο που είχαν είχε αυτή τη μορφή. Ήταν άειλο κεφάλαιο ουσιαστικά. Είχαν ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο ήταν απτό και το οποίο ήταν πολύ χαμηλής ποιότητας. Και ένα σημείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ αρνητικό στα πρότυπά μας είναι το γεγονός ότι είναι πολύ εύκολο να προσθέσει κανείς το goodwill, τη φήμη και την πελατεία στο, στον ισολογισμό μια τράπεζα ή μια, ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Νομίζω λοιπόν ότι εάν κάποιο είχε μια σωστή προσέγγιση θα είχε κατανοήσει ότι υπήρχε ένα πρόβλημα. Γιατί δεν έγιναν όμως αυτά πραγματικότητα, γιατί οι σταθμισμένοι λόγοι της ε, Βασιλείας επέτρεπαν στις τράπεζες να διακυβεύουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους και όταν είχαν εκθέσεις της τάξεως του 1000 παραδείγματος χάρη με τη στάθμιση κινδύνου θα φαινόταν ότι η έκθεσή τους ήταν μονάχα 300 και όχι 1000. Επομένως αρκούσε να βάλουν στην άκρη ένα μικρό ποσό ω κεφάλαιο ασφαλεία, ένα 10% παραδείγματο χάρη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βελτίωση σε σχέση με τους ε, λόγους ασφαλείας, τους κεφαλαιοχικούς λόγου τη Βασιλεία. Μπορείτε να με ρωτήσετε αν είναι επαρκέ αυτό και εγώ αναρωτιέμαι. Τουλάχιστον όμω γίνεται κάτι σε σχέση με τα προβλήματα αυτά και όπω σα είπα προηγουμένω, βελτιώνουμε και εμεί τα λογιστικά μα πρότυπα ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν και μελλοντικέ καταστάσει και όχι μόνο τωρινές καταστάσεις. Θα έπρεπε τώρα αυτά τα πρότυπα να οδηγούν τις τράπεζες στο να έχουν αποθέματα για απρόπτες απώλειες. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός ότι σε πολλές χώρες, σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιρλανδία, όπως είναι το... και άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι απώλειες στο σύστημα ήταν πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μπορούσε να προβλέψει ο οποιοδήποτε. Η Ισπανία είχε το σύστημα του Dynamic Provisioning, το οποίο υποχρέωνε τις τράπεζες να δημιουργούν ένα μαξιλαράκι για μελλοντικές ε, απώλειες. Έδωσε αυτό στις ε, Ισπανικές τράπεζες κάποιο περισσότερο περιθώριο. Αλλά αυτό το περιθώριο τελικά φάνηκε ότι ήταν απόλυτα ανεπαρκές για να καλύψει τις τεράστιες απόλυσεις που υπέστη το ισπανικό τραπεζικό σύστημα. Αν λοιπόν οι ίδιοι τραπεζίτες δεν μπορούν να προβλέψουν τις ε, απρόπτες απώλειες, αν το κάνουν αυτό δεν θα ήταν απρόπτες, αν δεν μπορούν να το κάνουν οι ρυθμιστικές αρχές, τότε μην περιμένετε τα λογιστικά πρότυπα να καλύψουν αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά δεν μπορεί κανεί να προβλέψει τι είναι απρόοπτο. Θα λέγαμε απλώ στου λογιστέ, βγάλτε ένα αριθμό από ένα καπέλο, βάλτε ένα οποιοδήποτε αριθμό θέλετε για απρόοπτε ε, και θα μας ε, περιγελούσαν οι αρμόδιοι στα χρηματοοικονομικά. Θα πρέπει όλοι να δούμε την ιστορία της, ε, χρηματοοικονομική, της χρηματοοικονομικής. Έχουμε κατά καιρούς κρίσεις και αν Υπάρχει ένα τομέας ο οποίος έχει σαν απόθεμα μόνο το 2-3% ε, του συνολικού κεφαλαίου. Ξέρετε ότι αυτό το 2-3% δεν μπορεί να καλύψει τις απρόπτες απώλειες. Έχουμε και άλλους οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Ναι, ναι, λέει ο Βολφ Κλίντς, είναι μια πολύ μικρή παρατήρηση. Μα δεν έχουν αποτύχει και οι ορκωτοί για τα θέματα αυτά. Μήπως θα έπρεπε να είχαν υποδείξει τον κίνδυνο αυτό εγκαίρως. Ναι, θα μπορούσαν να είναι πιο προορατικοί ίσως στις επαφές τους με τους ρυθμιστές. Για να σας πω όμως την αλήθεια, όσο λέγανε οι ρυθμιστικές αρχές όλα πάνε καλά, δεν είχαν κανένα κίνητρο να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου οι λογιστές. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιο επάγγελμα το οποίο δεν έχει διδαχθεί δεν έχει πάρει κάποια διδάγματα από αυτή την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Και οι λογιστές και οι τραπεζιτές και οι πολιτικοί χρειάστηκε να διδαχθούν αυτά τα πράγματα. Βέρνερ, μπορείς να, θες να επανέλθεις. Ναι. Ήθελα να, ρωτήσω ε, σε αυτό που αναφέρεται για την, το ιδιωτικό θέμα. Καλύτερα θα ήταν να είναι βέβαια στον ισολογισμό. Τώρα συμφωνήσαμε για το παράρτημα. Είναι τελική αυτή η απόφαση ή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Διότι μετά από ανακοίνωση του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου μετά από το 15 Οκτωβρίου 2008 1,27% των επισφαλών ε, αναφερόταν στους ισολογισμούς. 1,27% μόνο των επισφαλών ε, αξιογράφων και δανείων. Μπορείτε να μας πείτε τώρα τι γίνεται, ποια γραμμή ακολουθούν οι Αμερικανοί, προχωράν πολύ γρήγορα ή εθελοτυφλούν. it is, uh, uh, first of all... Να σας απαντήσω. Καταρχάς δεν προβλέπω μια νέα συμφωνία. Βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα πρέπει να το αποδεκτούμε τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Για ποιο λόγο τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε. Πολλά έχουν να κάνουν με το ότι στην Αμερικανική νομοθεσία υπήρχαν κάποιες, ε, κάποια κριτήρια όσον αφορά την μόχλευση, η οποία τα οποία κριτήρια είχαν περάσει σε κάποιους παλιούς λογιστικούς κανόνες. Και τα ποσοστά αυτά μόχλευσης βοήθησαν τελικά τις ΗΠΑ να κινηθούν καλύτερα μέσα στην οικονομική κρίση, καλύτερα σε σχέση με εμά. Πρέπει να ακολουθούμε άλλους λόγους, αυτούς που επιβάλλονται από τη Βασιλεία. Καθότι λοιπόν είχαν περάσει όλα αυτά τα κριτήρια στην Αμερικανική νομοθεσία, η ε, Κεντρική Αμερικανική Τράπεζα δεν ήθελε να αλλάξει σε εκείνη τη φάση τα λογιστικά πρότυπα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν τροποποιήθηκαν. Επομένω, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν παράτυπη η αντιμετώπιση του, αλλά θα ήταν σαφώ πολύ καλύτερα αν είχαμε ένα κοινό ενιαίο σύστημα. Εν γέννη πάντως μπορούμε να πούμε ότι ε, τα IFRS, τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, αποτελούν πρότυπα υψηλότερης ποιότητας σε σχέση με τα αμερικανικά. Εμείς καταφέρνουμε να πετύχουμε μια πολύ καλύτερη ομαδοποίηση, ένα πολύ καλύτερο συγκερασμό. Οι κανόνες που έχουμε για την ομαδοποίηση είναι πολύ πιο αυστηροί. Επομένως είναι πολύ δυσκολότερο στην Ευρώπη να κρατήσει κανείς πράγματα εκτός λογισμού, πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί πιο εύκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προερχόμενο από μια μεγάλη εταιρεία πληροφορικής όπου η μίσθος τελικά αποτελούσε ένα πολύ μεγάλο τμήμα των κερδών, συμφωνώ ότι η δήλωση των κερδών καθώς επίσης και η μίσθωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο του συλλογισμού. Είπατε ότι πολλές φορές η μίσθωση μένει εκτός. Πολλές φορές δεν δηλώνεται καθόλου. Υπάρχουν όμω και άλλοι θύλακε, αν θέλετε, στην οικονομία, όπου θα μπορούσαμε να είχαμε στοιχεία του παθητικού, τα οποία μένουν εκτός λογισμού τελικά και τα οποία θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και τα οποία θα έπρεπε εμεί να γνωρίζουμε. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερον, αναφερθήκατε σε κάποιες ε, απώλειες, σε κάποιες αναμενόμενε απώλειε. Δεν νομίζετε ότι ε, ενδεχομένως εμείς με τα πρότυπα αυτά να καταστήσουμε το όλο σύστημα πιο ασταθές ουσιαστικά να βρεθούμε μπροστά σε κάποιες καταστάσεις οποίες πραγματικά θέλουμε να αποφύγουμε. Νομίζω ότι ε, δεν είναι απόλυτη επιστήμη να καταφέρει κανείς να εκτιμήσει τις ε, απώλειες. Μήπως αν αρχίσουμε να εκτιμούμε και να καταγράφουμε τις ε, εκτιμόμενες απώλειες, μήπως αυτό λειτουργήσει τελικά σαν μπούμεραγκ. Αναφερθήκατε επίση στα κριτήρια της Βασιλείας και αναφερθήκατε στις κρηματοοικονομικές αναφορές ανά χώρα. Είπατε ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν. Η Επιτροπή της Βασιλείας όμως είναι ένας οργανισμός που παρτίζεται από ρυθμιστικές αρχές και από τους επικεφαλείς των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών. Πρόκειται για δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν νομοθετούν αλλά προτείνουν κανόνες. Επομένως, εγώ συμφωνώ ουσιαστικά με αυτούς οι οποίοι λένε ότι ο δικός σας οργανισμός δεν έχει το απαραίτητο επίπεδο λογοδοσίας προκειμένου να καταρτίζει κανόνες. Τα κοινά λογιστικά πρότυπα αποτελούν ένα κοινό αγαθό. Πώς μπορούμε εμείς να ιδιωτικοποιήσουμε τελικά την κατάρτιση των προτύπων αυτών σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν λογοδοτούν. και φοβάμαι πολλές φορές ότι ε, ακριβώς επειδή ορισμένε μονομένες χώρες δεν συμφωνούν με τις δικές σας προτάσεις, μπορούμε τελικά να μην καταλήξουμε σε αυτά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στην ευρύτερη εμβέλειά τους. Κοιτάξτε, κάνουμε πολλά πράγματα που με τα οποία πολλοί δεν συμφωνούν, όπως για παράδειγμα το κριτήριο αυτό, το πρότυπο αυτό που έχει να κάνει με τη μίσθωση. Κοιτάξτε, η δική μας οργάνωση πραγματικά είναι αφοσιωμένη στο κοινό καλό. Ο Επίτροπο Μπαρνιέ ήρθε στα γραφεία μα πριν από μερικού μήνε και πραγματικά εντυπωσιάστηκε από τη φιλοδοξία των εργαζομένων μα ότι πραγματικά είναι ταγμένοι στο κοινό καλό. Και ναι, όντω καταρτίζουμε κανόνε, αλλά εσεί τελικά αποφασίζετε για το αν θα εφαρμοστούν οι κανόνε αυτοί ή όχι. Πρόκειται για μία απόφαση που κοινοβουλευτικά λαμβάνεται στα περισσότερα κράτη-μέλη. Ορισμένα μόνο κράτη-μέλη έχουν ε, εντάξει στην νομοθεσία τους Μία ρήτρα η οποία λέει ότι οι δικές μας οι οδηγίες αποτελούν αυτόματα νομοθεσία. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει μια διαφορετική κοινοβουλευτική εσωτερική διαδικασία η οποία μπορεί να εγκρίνει ή να τα απορρίψει τελικά τις δικές μας τις οδηγίες. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των κανόνων μας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κάθε χώρα αρχίσει να τροποποιεί εν μέρη τις δικές μας τις οδηγίες, δεν θα καταλήξουμε ποτέ σε ενιαία λογιστικά πρότυπα. Προφανώς όμως έχετε μια απόλυτη εθνική κυριαρχία και εσείς τελικά αποφασίζετε για το αν θα εφαρμόσετε ή όχι τα λογιστικά μας πρότυπα. Η δημόσια λογοδοσία μας πραγματικά έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ιδίως με την σύσταση του Monitoring Board, του Συμβουλίου αυτού εποπτείας, στο οποίο συμμετέχουν και οι διαχειριστές μας. Επομένως, έχει ενισχυθεί η δημόσια λογοδοσία μας και θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Και ως πρώην πολιτικός, ειλικρινά σας λέω, ότι μ' αρέσει η εξέλιξη αυτή. Market-to-market -market accounting. Ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πολύ συχνά και ξέρετε ότι πάρα πολλοί παραπονιούνται τελικά όταν οι τιμές αυξομειώνονται. Καταρχάς, εμείς δεν προωθούμε στα πλαίσια του δικού μας οργανισμού το market-to-market -market accounting. Χρησιμοποιούμε διαφορετικά συστήματα, ένα συνδυασμό διαφορετικών συστημάτων και δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα κριτήρια. Και ξέρετε ότι θέλουμε να έχουμε μια πολύ διαφορετική, διαφοροποιημένη αντιμετώπιση όσον αφορά τις, τα κρατικά ομόλογα. Διαφορετική στάση έχουν προτείνει οι Αμερικάνοι, οι οποίοι θέλανε να υπήρχε μια κοινή τιμή. Εμείς θεωρήσαμε ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, σε μια αποτίμηση σε συνθήκες αγοράς. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, μια τράπεζα, η Deutsche Bank, χρησιμοποίησε διάφορα τοξικά μέσα, όπως ε, μέσα τα οποία χρησιμοποιούσαν ακριβώς αυτό το market-to-market -market accountability. Στον δικό του ισολογισμό, στον ισολογισμό της τράπεζας αυτής υπήρξε μια πολύ απότομη μείωση των τιμών Κατάφεραν όμως εγκαίρως να αποκλείσουν από τον ισολογισμό τους αυτά τα τοξικά μέσα και κατάφεραν ουσιαστικά να κρατήσουν ένα πιο υγιή ισολογισμό. Η αξία των μέσων αυτών δεν επηρεάστηκε άμεσα από την αξία που υπήρχε στην αγορά Επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ θετικό να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην αγορά και νομίζω ότι μια τράπεζη η οποία δεν παρακολουθεί την αξία που έχουν στην αγορά τα μέσα στα οποία επενδύει, αυτόν μη τι άλλο αποτελεί μια πολύ ανεύθυνη στάση. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Ε, οι συντάξει, παραδείγματο χάρη, οι συντάξει ήταν εκτό ισολογισμού για πολύ καιρό. Και τώρα πολλά ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω του μηδενικού επιτοκίου που λαμβάνουν από τις επενδύσεις τους και της οικονομικής κρίσης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για τον επενδυτή να ξέρει τι παρουσιάζεται. Όταν προτείναμε το συνταξιοδοτικό ή το κόστος των συντάξεων να υπάρχει στον ισολογισμό, πάρα πολλές εταιρείε δεν ξέρανε ακριβώς τι είναι αυτό το ποσό και για πρώτη φορά εξαναγκάστηκαν να κάνουν ακριβείς υπολογισμού του παθητικού τους για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ναι, το leasing, οι χρονομερισματικές μισθώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που ξέρουμε ότι έχει ξεφύγει από μας, ε, μας έχει διαφύγει. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένα κενά, ορισμένα, ορισμένες ελλείψεις, αλλά εγώ είμαι, δεν αισθάνομαι πολύ άνετα με το θέμα του goodwill, της υπεραξίας. That is something I'm worried Τη φήμη και πελατεία. ναι, το οποίο πολλέ φορέ δεν είναι στο μισολογισμό Η πρόεδρος. Λοιπόν, ας ε, συνεχίσουμε με το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που για την επίσκεψή σας, ο κύριος Γκίγκολτ. Έχω ένα ερώτημα το οποίο αφορά την εσωτερική σας, τον εσωτερικό σας κανονισμό λειτουργίας. Μέχρι τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο ανανενόταν από μόνο του. Αυτό δημιούργησε πολλές επικρίσεις, αυτή η μέθοδος δηλαδή αυτοανακύκλωσης και είπατε και εσείς ο ίδιος ότι υπάρχει μια εποπτική αρχή πλέον, ένα monitoring board που λειτουργεί. Όμως εγώ πιστεύω ότι το δημοκρατικό έλλειμμα υπάρχει ακόμα στον οργανισμό σας. Θα ήθελα να ξέρω ακριβώς τι λειτουργίες έχει αναλάβει το Εποπτικό Συμβούλιο, πώς εκλέγονται τα μέλη και τι γίνεται με τη διαφάνεια της εσωτερικής σας λειτουργίας, δηλαδή του τρόπου λειτουργίας σας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και τις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου ο, ο κύριος Χόγκερφορστ. Θα ήθελα να πω ότι μετά από μια μακρά καριέρα στην πολιτική και σε στο κανονιστικό πλαίσιο, ποτέ δεν έχω εργαστεί σε ένα περιβάλλον με τόση πολύ διαφάνεια. Όλα γίνονται δημόσια. δεν υπάρχει δυνατότητα, απαγορεύεται σε εμά να κάνουμε συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών. Δεν μπορούμε να μαγειρέψουμε ή να προετοιμάσουμε, να προαποφασίσουμε τις συνεδριάσεις μας, διότι είναι δημόσιες. Όποιος θέλει μπορεί να τις παρακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχει πραγματικά ε, απόλυτη ε, εποπτεία και έλεγχος αυτών που λέμε και κάνουμε. Είμαστε, κάθε φορά που παίρνουμε μία απόφαση γίνεται μία συνεδρίαση και για τα πρακτικά υπάρχει ένα ε, χρονικό περιθώριο 120 ημερών για αντιρρήσεις, να υποβληθούν αντιρρήσεις για τροποποιήσεις και σχόλια η αρνητική πλευρά όλης αυτής της διαφάνειας και της δημοσιότητας είναι ότι καθυστερούμε πάρα πολύ να καταλήξουμε σε μία απόφαση. Ε, πολλές φορές έλεγα ότι οι πολιτικοί καθυστερούν πολύ στη λήψη των απεφάσεων. Πολλές φορές για ένα πρότυπο, ένα διεθνές πρότυπο, χρειαζόμαστε πέντε ή δέκα χρόνια το διοικητικό μας συμβούλιο ελέγχεται από το εποπτικό συμβούλιο. Το εποπτικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ε, και με συνένεση ε, και εγκρίνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πάλι οι συνεδριάσεις του είναι ανοιχτές, είναι δημόσιες. Είμαστε υπόλογοι. Είμαστε υπόλογοι έναντι αυτού του Διεθνούς Συμβουλευτικού Φορέα ε, και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερη η καταγραφή των απόψεων των ε, ε, Ευρωπαίων και των υπερατλαντικών μας εταίρων. Ε, παραδείγματος χάρη στο Διοικητικό Συμβούλιο του συμβουλευτικού φορέα θέλουμε ε, ε, να εκλεγεί κάποιος, η ΙΦΡΑΚ ε, ελέγχει με μεγάλη ακρίβεια τι προσπάθειες έχουμε κάνει για την επικύρωση και υιοθέτηση του ενός ή του άλλου προτύπου. Μπορεί να μας επικρίνει, να σχολιάσει αυτά τα οποία έχουμε κάνει, να μην συμφωνεί με κάτι το οποίο έχουμε κάνει. Αλλά εμείς, δεδομένου ότι θέλουμε να ενεργούμε πάντοτε πρακτικά, πρέπει να ακούμε, πρέπει να ακούμε την άποψη τους. Η, η Βασιλεία, η, Επιτροπή τη της Βασιλείας μπορεί να είναι ε, δημόσια, αλλά οι συνεδριάσεις τους δεν είναι. Δεν είναι, δεν υπάρχει διαφάνεια στις συνεδριάσεις τους. Άλλο τι γίνεται μετά. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω και να σχολιάσω περιττέρω. Σέβομαι ιδιαίτερα τους συναδέλφους μου που συμμετέχουν στην Επιτροπή Βασιλείας, αλλά δεν είναι όσο διαφανής εμείς. Ο κύριος Γκίγκολτ, θα ήθελα να ξέρω πού καταγράφονται οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, πού καταγράφονται και πού μπορώ να βρω τις αποφάσεις αυτές, ποιος και ποιος συμμετείχε στην λήψη των αποφάσεων υπάρχει ε, πάντοτε μία δήλωση ε, μετά από τη συνεδρίαση του Ποπτικού Συμβουλίου και μέρος της συνεδρίασης είναι δημόσιο και, δημοσι... και δημοσιεύεται και online. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος, η πρόεδρος. Ε, δεν πρέπει ακόμα να φύγετε. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Ωραία, σας κρατάμε όμοιρο λοιπόν για λίγο ακόμα, γιατί υπάρχουν ακόμα ορισμένα μέλη μας που πρέπει που θέλουν κάτι να ρωτήσουν και είμαι και εγώ στον κατάλογο των ομιλητών. Ήμουν πολύ υπομονετική μέχρι τώρα. Ξέρετε ότι εδώ και πολύ καιρό με έκαιγε ένα θέμα ε, της ρευστότητας, ε, του cash flow και βασικά δεν μου αρέσει το στοιχείο αυτό είτε υπάρχει στον ισολογισμό είτε στους ε, ε, λογαριασμούς που παρουσιάζονται ε, και εν μέρει έχετε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα ιδίω όσον αφορά εκεί που υπάρχει διαφορές, διαφορά μεταξύ του, των αποσβέσεων και του, της, του cash flow, της ρευστότητας. Ε, ορισμένες φορές τα στοιχεία αυτά δεν υπήρχαν καθόλου ε, στους ε, ισολογισμούς. Τώρα μπορούμε τουλάχιστον να ανοιχνεύσουμε ορισμένα στοιχεία. Τώρα, εάν οι ζημίες ξεπεράσουν τις προσδοκίες ή αυτά που υπολογίζαμε, είχαμε και το πρόβλημα αυτό στο παρελθόν. Υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση στην αναγνώριση αυτού του γεγονότος. Τι έχετε κάνει για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Uh, going from Δεδομένου ότι πρέπει θέλουμε υποτίθεται να είμαστε ουδέτεροι στους κανονισμούς ε, από την ε, ίσως ε, υπερβολική μετριοφροσύνη και, και να πάμε στην ουδετερότητα. Αλλά τι, τι ωφελεί η ουδετερότητα όταν πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Και τι, τι γνώμη έχετε για το ρυθμιστικό hedging, δηλαδή την ε, πρόληψη κινδύνων και την ε, προστασία έναντι μελλοντικών κινδύνων και την ε, τι συναλλαγέ αυτού του τύπου, του hedging. Παραδείγματο χάρη μια τράπεζα εκδίδει αξιόγραφα ή έχει αξιόγραφα και εν συνεχεία κατακρατεί το 20% έναντι της συνολικής αξίας και εν συνεχεία κατακρατεί και άλλα 10% και αυτή η αναλογία 20 με 50% οπότε αντί για 20% που είπε κρατάει 10% για ασφάλεια Οπότε το, το CDS δεν θα υλοποιηθεί ποτέ, διότι θα κρατηθεί αυτό το απόθαμε έναντι μελλοντικών συναλλαγών. Έχουμε λοιπόν ένα hedging, ένα, μία εξαγορά των, των αξιογράφων αυτών ε, του ύψους του 10% ε, το οποίο δεν διατίθεται είναι μία προσκομματική διαδικασία αυτή. Πώς νομίζετε ότι επιβεβαιώνεται η αξία αυτής της δυνατότητας που έχουν οι τράπεζες να το κάνουν. Ο, ο κ. Σούγκες πρόκειται. Καταρχάς, εμείς δεν είμαστε ρυθμιστές, δεν κάνουμε κανονιστική εργασία, εμείς εκδίδουμε ε, λογιστικά πρότυπα. Και ο στόχος μας δεν είναι να επιβάλλουμε κανόνες στις τράπεζες ή σε εταιρείε για το πώς θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Ε, εμείς θέλουμε να τους δείξουμε τι έγινε στο παρελθόν και το να μπορούμε να τους πείσουμε και τους δείξουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι κάποιος είπε ακριβώ ότι η λογιστική είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη. Πράγματι, η, αλήθεια δεν, δεν ε, απέχει και πολύ από αυτή τη δήλωση. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της, yeah. um... της σύνεσης, η ουδετερότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν είσαστε υπερβολικά συντηρητικοί στα λογιστικά σας, υπερβολικά συντηρητική και αυτό έγινε στο παρελθόν όπου οι τράπεζες και οι εταιρείε μπορούσαν να, να έχουν τον κουμπαρά γεμάτο έτσι ώστε στις κακές εποχές να μπορούν να, να τραβάν κονδύλια. Ε, εντάξει, αυτό ήταν πάρα πολύ ασφαλές κατά κάποιον τρόπο, αλλά αυτό το οποίο εχθές ήταν συντηρητικό, ε, αύριο αλλάζει φύση όταν η απόδοσή σου αρχίζει και γίνεται αρνητική, φθήνει, ο επενδυτής δεν βλέπει τη χειροτέρευση, αλλά βλέπει μια σταθερή ροή και δεν βλέπει, δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι η τράπεζα φθήνει, παίρνει έναν κατήφορο. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι η δοτερότητα έχει εξαιρετική σημασία έτσι ώστε ο ισολογισμός κερδών και ζημιών να μπορεί να αντανακλά ε, την πορεία μιας τράπεζας ή μιας εταιρείας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε πολλά πρότυπα δεν εφαρμόζουμε την σύνεση. Ξέρουμε ότι τα, λογιστικά, η λογιστική ε, επιστήμη δεν είναι ε, τόσο επακριβής όσο 100% ας πούμε, αλλά προσπαθούμε να συνυπολογίσουμε και μία θεμητή αξία. Πολλές φορές δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε μία αξία, ούτε να προβλέψουμε, ας πούμε, ακριβώς το χρηματοοικονομικό, την επίπτωση του χρηματοοικονού προϊόντος. Γι' αυτό προσπαθούμε στις εκθέσεις και στους ελέγχους να, να τονίσουμε ποια είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιο είναι το ρίσκο ιδίως σε ένα spread, σε μια ας πούμε, οριζόντια διαδικασία της τράπεζας. Και στο μοντέλο υπολογισμού, προληπτικού υπολογισμού απολειών, ζημιών, προσπαθούμε να αποφύγουμε μια υπερβολικά αισιόδοξη εικόνα. Και αυτό το ερώτημα έχει ζητηθεί και στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου και η Βρετανική κυβέρνηση είπε ότι είχε είχε το, το, το αίσθημα ότι η συνένεση είναι ακόμα μια κατευθυντήρια γραμμή του IFRS και συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχει ακόμα το στοιχείο της σύνεσης. Πρόσφατα ε, έκανα μια ομιλία που υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας περί σύνεσης και έδωσα αρκετά παραδείγματα για το πού ακόμα εφαρμόζεται αυτή η σύνεση, αυτή η προσοχή ας πούμε, που προσδίδουμε. Μπορείτε να τα δείτε αυτά στην ιστοσελίδα. Καιρός να σταματήσουμε, ναι πράγματι. Εννοείται. Τι εννοείται. Όπως είπα και προηγουμένως, οι περισσότερες τράπεζες βρίσκονται κάτω από την ε, εύλογη αξία τους αυτή στο χρηματιστήριο, η αξία τους στο χρηματιστήριο. Πολλές από αυτές βασίζονται ακόμα στην θύμη και την πελατεία. Αναρωτιέμαι αν είναι αρκετά αυστηρά τα πρότυπά μας, ώστε να μπορούν τράπεζες οι οποίες βρίσκονται σε τόσο δύσκολη κατάσταση χρηματοπιστωτικά να εμφανίζουν φήμη ή πελατεία στη, στους ισολογισμούς τους. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αλλά κάτι το οποίο δεν με κάνει να νιώθω πολύ άνετα. Θεωρείτε ότι όταν υπάρχει μια συγχώνευση ε, επιχειρήσεων θα πρέπει να απομειώνεται η φήμη και πελατεία, όπως γινόταν, έτσι γινόταν στο παρελθόν. Κανονικά υπήρχε μια διαδικασία απόσβαση σε 20 χρόνια. Και αυτό έχει ένα χαρακτήρα αυτερεσία. Δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε ένα τέτοιο κανόνα. Όταν γίνεται μια συγχώνευση επιχειρήσεων και περιμένει κανεί να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των δύο επιχειρήσεων και αυτό πληρώνει κανεί περισσότερο πάνω από την χρηματιστική αξία μια εταιρεία. Θα ήταν λογικό αυτές οι συνέργειες να οδηγήσουν και σε μια απομείωση στον ισολογισμό μέσα στα επόμενα ας πούμε 7 χρόνια. Και δεν είμαι σίγουρος αν συμβαίνει αυτό πάντα στην πραγματικότητα. Ωραία. Ε, ο κύριος Κεμάλ και πάλι. Επανέρχομαι στο θέμα των συγχωνεύσεων. Όταν ήμουν στον ακαδημαϊκό τομέα, κάτι το οποίο έλεγα πάντα στους φοιτητέ μου είναι ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο έχει νόημα ε, δύο εταιρείε να συγχωνεύονται είναι οι συνέργειες. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συγχωνευτούν. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι η άποψη που διατύπωσα ότι ορισμένοι θεωρούν ότι η ερμηνεία του true and fair, δηλαδή ότι απεικονίζουν τα λογιστικά στοιχεία την κατάσταση μιας επιχείρησης, ότι θα πρέπει πράγματι να είναι αυτό που διέπει τους λογαριασμούς. Αυτά τα οποία λέει η IFRS έχουν μια τελείως διαφορετική ερμηνεία από αυτά που βρίσκονται στην τέταρτη και έβδομη οδηγία για τα εταιρικά θέματα. Επομένως, ουσιαστικά παραβιάζουν αυτά τα πρότυπα την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν μια παρατήρησή μου. Και δεύτερον, η διάκριση μεταξύ ε, προβλεπτών και απρόβλεπτων ε, ζημιών είναι πολύ δύσκολη. Αλλά αν έχει κανείς ήδη ένα αποθεματικό για ε, απώλειες, τότε θα πρέπει κανείς να ξέρει ακριβώς πόσο μεγάλες είναι οι υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν, το παθητικό που μπορεί να προκύψει. Είδαμε λοιπόν στην κρίση τι γίνεται, ότι όταν τα πράγματα πήγαιναν στραβά, κανείς δεν είχε τον τρόπο να υπολογίσει το, την προσδοκόμενη απώλεια με ένα μοντέλο. Δεν μπορώ να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Για το δεύτερο ερώτημα, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό. Ελληνιστή CDS λέμε. CDS λέμε και στα ελληνικά. Ε, στο αμερικάνικο σύστημα. Θέλει κανείς να δημιουργήσει ένα σύστημα ώστε όταν συνάπτει ένα δάνειο ήδη προβλέπει ποια είναι η ε, δυνητική απώλεια από αυτό το δάνειο και επομένως γίνεται μια απόσβεση με τη βάση αυτή. Και πάλι όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Γιατί η τιμή πρόσκτησης ενός δανείου μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερη από την τιμή αγοράς. Και έτσι δεν δείχνουμε την τιμή, την τιμή της αγοράς πράγματι. Αυτό είναι αρνητικό. Επίσης υπάρχουν παράπλευρες συνέπειες που μπορούν να προκύψουν όταν έχουμε δάνεια στα οποία οι προσδοκόμενες απόλυσεις είναι οι πιο υψηλές, είναι ουσιαστικά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δάνεια όπου οι τράπεζες ζητούν μεγαλύτερη ψαλίδα επιτοκίων για να καλύψουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, γιατί είναι δάνεια τα οποία δεν είναι επενδυτικού χαρακτήρα. Αν μια τράπεζα πρέπει να ξεγράψει τελείως αυτά τα δάνεια όταν τα δίνει και να τα απομειώσει στα λογιστικά του. στοιχεία, τι θα γίνει σε μια κρίση όπως η σημερινή, όπου είναι ήδη πολύ μικρός ο αριθμό των δανείων προ μικρομεσαίε επιχειρήσει, θα σταματούσαν να δανείζουν μικρομεσαίε επιχειρήσει, γιατί αυτό θα έπλητε τα, την κερδοφορία του. Θα δείχνανε καλύτερα στοιχεία ε, ισολογιστικά εάν δεν κάναν καθόλου δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν λοιπόν και συνέπειες οι οποίες μπορούν να προκύψουν και οι οποίες θα ήταν αρνητικές και δεν θέλαμε να τις προκαλέσουμε. Θεωρούμε ότι δεν ήταν καλύτερο να εξασφαλίσουμε ότι μία τράπεζα δεν θα πρέπει να αναγνωρίζει όλη την κερδοφορία που έχει σε επισφαλή δάνεια. Να μην λοιπόν καταγράφει όλα αυτά ως κερδοφορία όταν είναι καλά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρει αν τελικά θα μπορέσει να πάρει πίσω τα, τα δάνεια αυτά. Και όταν ξέρει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πλήρης ε, αποπληρωμή των ε, δανείων, μόνο τότε να καταγράφεται η ζημία. Όσο όμως τα δάνεια δίνουν, εξυπηρετούνται, τότε το κέρδος των δανείων δεν θα πρέπει να αντανακλά το πριν κινδύνου, αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να απομειώνονται σε σχέση με το πριν κινδύνου που έχει να κάνει με το πόσο επισφαλή είναι αυτά τα δάνεια. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε κάτι το οποίο έχει οικονομική λογική. Οι τράπεζες μας λένε δεν μπορούν να λειτουργήσουν με βάση με ένα τέτοιο μοντέλο και τα πράγματα τα οποία μπορούν να απεικονίσουν λειτουργικά, πολλές φορές αυτό δεν έχουν και οικονομικό, οικονομική λογική πίσω τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Είπατε προηγουμένως, λέει ο Βένερ, ότι δεν συμφωνείτε με όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. Υπάρχει μια απόφαση η οποία ελήφθη μέσα στην κρίση χρέους ότι στο μέλλον τα κρατικά ομόλογα ανεξάρτητα από που ε, υπήρχε μάλλον η απόφαση όλα τα κρατικά ομόλογα να έχουν μηδενική στάθμιση κινδύνου. Συμφωνείτε με κάτι τέτοιο. Μήπως σε κάποιο δεκα διάστημα μετα, ε, μεταβατικό θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα αυτά. Θεωρείτε ότι μπορεί τη στιγμή που δεν είναι η ίδια η αξιοπιστία όλων των κρατικών ομολόγων να έχουν όλα μηδενικό, ε, μηδενική στάθμιση κινδύνου. Όταν το ρωτάτε το ερώτημα με αυτόν τον τρόπο, το έχετε απαντήσει ήδη. Δεν είμαι ρυθμιστή για τα τραπεζικά θέματα. Νομίζω ότι η Επιτροπή της Βασιλείας έχει κάνει πολύ καλό έργο. Αλλά σίγουρα αυτό είναι και το μαλακό υπογάστριο, αν θέλετε, τη ρυθμιστής Βασιλείας. Κοιτάξτε την περίπτωση τη Ιρλανδία. Η Ιρλανδία πριν από την τραπεζική κρίση είχε χρέο κρατικό 20% του ΑΕΠ, που ήταν το χαμηλότερο τη Ευρώπη, Με την κρίση μετά από δύο χρόνια ξεπέρασε το 120 του ΑΕΠ και ουσιαστικά μειώθηκε σε επίπεδο junk η αποτίμηση αυτού του χρέους. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα απόλυτα ασφαλές στοιχείο ενεργητικού. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν υπήρξαν απόλυτα ε, ασφαλείς επενδύσεις ή ασφαλή στοιχεία ενεργητικού. Ακόμα και χώρες σαν η Γερμανία ή οι κάτω χώρες, η χώρα μου, που φαίνεται ότι βρίσκονται ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση και εμεί ακόμα έχουμε πληγεί από αυτή την κρίση και κανεί δεν ξέρει τι θα προκύψει τελικά. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα ασφαλή, 100% ασφαλή. Γι' αυτό θεωρώ ότι η μηδενική στάθμιση στο κρατικό χρέο σίγουρα δεν αντανακλά τι οικονομικέ πραγματικότητε. καλά. Κάποιος άλλος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε πέρα από το χρόνο που προβλεπόταν και ελπίζουμε να σας έχουμε και πάλι μαζί μας στο ορατό μέλλον. Σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Thank you. Um, I'm now, uh, Ευχαριστούμε λοιπόν. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη στη συνέχεια. κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα καταρχάς. Right, so the next item is not going to happen until 5.30. Uh, Στις 5.30 uh, θα ασχοληθούμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έκθεση για την ανταγωνιστικότητα. Δεν θα καλύψουμε λοιπόν την έκθεση του κυρίου Στόλογιαν, γιατί δεν είναι εδώ, δεν είναι διαθέσιμος. Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με την έκθεση αυτή, αλλά δεν είναι η Σόρφιν Βέλτ εδώ ούτε οι υπόλοιποι συνεργάτες του κυρίου Στόλογεν. Λυπάμαι που θα σας ζητήσω να ξανάρθετε εδώ στις 5.30 σήμερα. Κάνουμε διάλειμμα λοιπόν για μία ώρα και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την έκθεση ανταγωνιστικότητας. δεν βλέπω Okay. Ωραία. Αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να ξαναρχίσουμε με το θέμα 6. Ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν η πολύ ενδιαφέρουσα ισπανική διμερή συζήτηση ολοκληρωθεί, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Αντολή, να έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μια συζήτηση για τις τροπολογίες που αναφέρονται στην έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Νομίζω ότι μπορώ να σταθώ πολύ σύντομος, γιατί ο ρόλος μου θα έπρεπε να είναι να δώσω απάντηση στα σχόλια αυτών που έχουν καταθέσει τροπολογίες. Ίσως μπορώ να πω κάποια πράγματα για την ε, μορφή της έκθεσης. Είχε 24 αιτιολογικές σκέψεις, 3 αιτιολογικές αναφορές και 24 εκτελεστικά στοιχεία, 150 τροπολογίες περίπου, μερικές από τις οποίες είναι δικές μου. Εγώ είχα σαν στόχο να συμπληρώσω αυτή την ετήσια έκθεση. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες από τον κύριο Γκαρίγα που αναφέρονται κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι κρατικές επιδοτήσεις έχουν τεθεί υπό έλεγχο και το θέμα είναι το θέμα της ανάκτησης των κονδυλίων αν θεωρηθούν ότι δεν ήταν θεμητές. Αν είναι η καλύτερη λύση η ανάκτηση των ποσών αυτών ή αν μπορούν να υπάρξουν ε, αντι, εναλλακτικές ε, ρυθμίσεις και θεραπείες οι οποίες θα επαναφέρουν το θεμητό ανταγωνισμό αλλά δεν θα έχουν τόσο αρνητικό αποτέλεσμα σε επίπεδο χάρη απασχόλησης. Δηλαδή να έχουμε μια πιο ευφυή εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού. Άλλη τροπολογία που έχω καταθέσει αναφέρεται σε ορισμένε περιπτώσει όπου από τα κράτη-μέλη, όταν έχουν υπάρξει αθέμητε ανταγωνιστικέ πολιτικέ, ιδίω σε τομέα χρηματοπιστωτικό, να εξασφαλίσουν την επαναφορά τη νομιμότητα και τη ομαλότητα. Όταν γίνονται λοιπόν προσπάθειες για να επαναφερθεί η πραγματικότητα, η σωστή θεμητή κατάσταση, αυτές οι ενέργειες δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν κρατικές επιδοτήσεις γιατί δεν δίνουν σε κανένα ένα πλεονέκτημα, απλώς επαναφέρουν την πρώτερη κατάσταση και νομίζουμε ότι μπορούμε να θεωρήσουμε πράγματι ότι είναι θεμητές αυτές οι ενέργειες που έχουν σαν αποτέλεσμα να επαναφέρουν την πρώτερη κατάσταση κατά Δεν έχω παρουσιάσει άλλες τροπολογίες θα ήθελα να απαντήσω εάν κάποιος θέλει να αναφερθεί σε κάποιες τροπολογίες και φυσικά εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάλει στην βελτίωση αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τροπολογιών, αλλά ευτυχώς δεν είναι υπερβολικός και μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβατικές λύσεις. Ο Γκούναρ Χέρκμερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εισηγησή του Τρία σημεία είναι σημαντικά για να τα παρακολουθούμε στις μελλοντικέ εργασίες. Πρώτον, αυτό που τονίζεται και στην έκθεση είναι η σημασία και οι επιπτώσεις στην οικονομία ε, λόγω ενός καλού θεμητού ανταγωνισμού, ιδίως στον τομέα των τροφίμων όπου περισσότερος ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για τους πολίτες μας. Το ίδιο ισχύει βεβαίω και για άλλους τομείς της οικονομίας. Και είναι σημαντικό να παρακολουθούμε αυτήν την πορεία έτσι όπως θα την παρουσιάζει ο εισηγητής και έρχομαι στο δεύτερο ε, κέριο σημείο. Είναι ουσιαστικό να εξασφαλίσουμε το άνοιγμα στον ανταγωνισμό και στα κράτη-μέλη. Έχω ορισμένε τροπολογίες όσον αφορά τις υπηρεσίε γενικής φύσεως που όπως ξέρετε έχει, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των οικοκυριών και των πολιτών μας. Και ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών μας υπηρεσιών ε, παράγεται εκεί ακριβώς και είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε ε, τους ε, δημιουργούς, τους παραγωγούς αυτών των υπηρεσιών, αλλά και να ε, ενσαρρύνουμε, να επιδοτούμε τις ευκαιρίες των πολιτών να συμμετάσχουν σε αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να υπάρχει πλουραλισμός και επαρκές επιλογές διότι εδώ μιλάμε για τα χρήματα των φορολογούμενων και τα χρήματα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση ε, της ζωής των πολιτών μας, όχι μόνο δηλαδή στη στήριξη των παραγωγών αυτών που δημιουργούν τις υπηρεσίες. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα στην Επιτροπή εδώ η τρίτη που ε, παρατήρηση αφορά στην νομιμότητα, στην νομική ισχύ. Βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να, είναι, να συνάδουν και να είναι συμβατά με την νομοθεσία. Το πιο σημαντικό όμως πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην προσπαθήσουμε να απαλύνουμε τη γραφειοκρατία με αυτόν τον τρόπο, διότι είναι σαφές ότι έχουμε σαφή κριτήρια για το πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κρατικές ενισχύσεις. Δεν πρέπει πάση θυσία εμείς να ενσαρρύνουμε τις κρατικές ενισχύσεις παντού και πάντοτε πρέπει να προσέξουμε να αποφύγουμε τις τρευλώσεις του ανταγωνισμού, να μην αποθαρρύνουμε νέους ανταγωνιστές και θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Πότε μπορούμε να δώσουμε κρατική ενίσχυση, αλλά και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δίνοντας αυτή την κρατική ενίσχυση η επίπτωση είναι πρόσθετη αξία, προστιθέμενη αξία για τους χρήστες, για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Σόφη δεν είναι εδώ. Και χάσαμε και τον Φιλίπ. Οπότε δίνω το λόγο στον... Thank you, Mrs. Σας ευχαριστώ κύριε Σας ευχαριστώ. Σας Πρόεδρε. Διάβασα την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις από τις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσα. Θα σας πω για ποιο λόγο επίσης είναι σημαντικές. Καταρχάς, παράγραφος 3, όπου αναφερόμαστε στην επιτυχή εφαρμογή υλοποίηση του καθεστώτος αντιμετώπισης της κρίσης. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό στο παρελθόν, το ξαναλέω, ότι τα μέτρα αυτά είναι συνήθως προσωρινά. Δύο εκθέσεις έχουν υποβληθεί, στις οποίες αναφέρεται στο ζήτημα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Για τρίτη φορά λοιπόν επιμένω στο σημείο αυτό. Αναγνωρίζω βέβαια την εργασία που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα αυτό, ωστόσο θεωρώ ότι θα πρέπει να τους πιέσουμε να ακολουθήσουν την περιγραφόμενη διαδικασία το στομότερο δυνατό. Απότερο στόχος της πολιτικής ανταγωνισμού είναι να καταρριφθούν όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, προϊόντων, υπηρεσιών, αγαθών. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να αποτελεί ένα ουδέτερο μηχανισμό στα χέρια ουδέτερων παραγόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μην συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι πολιτικοί στόχοι, δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αυτή. Τρίτον, σε σχέση με αυτό θα μιλήσω για τις υπηρεσίες κοινή ωφελίας. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση να εξερθούν ορισμένες υπηρεσίες χωρίς να προβλέπεται κανένα κατόφλι. Ακόμα και αν υπάρχει ένα ελάχιστο κατόφλι πάλι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κίνδυνος καθότι μπορεί πάρα πολλοί πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών να εξαιρεθούν από τον έλεγχο των αρμόδιων εθνικών αρχών. Ο έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών και προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να μην καταβάλουν ένα πολύ ψηλό τίμημα για τις υπηρεσίες αυτές. Ελπίζω η έκθεση αυτή πραγματικά να επικεντρωθεί στο βασικό της στόχο και να μην επικεντρωθεί σε ζητήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσουμε την υλοποίηση πολιτική ανταγωνισμού στο δυνατόν περισσότερο. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Γιώργιν. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ευθύ εξ αρχή ότι δεν είμαι διόλου κατά τον ανταγωνισμό όπως πολλές φορές ε, κατηγορούν τους αριστερούς Έχω όμως ορισμένες επιφυλάξεις. Ε, συμφωνώ με τον Γκούναρ ότι ο ανταγωνισμός χρειάζεται για να αποφύγουμε τα μονοπόλια. Όμως ε, δεν συμφωνώ και με όλες τις απόψεις του Γκούναρ που λέει ότι η ζωή των πολιτών μας έχει βελτιωθεί, ότι μόνο βελτίωση έχει υπάρξει μέσω του ανταγωνισμού. Εγώ νομίζω ότι η απλούστευση της ζωής των πολιτών μας είναι πιο σημαντική. Ε, βέβαια και η παραγωγή, ας πούμε αυτοί που δημιουργούν τα προϊόντα, τις υπηρεσίε και αυτοί οι άνθρωποι, οι πολίτες είναι. Άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των μεν και των δε. Ε, στην Ομοσπονδιακή Γερμανία δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί θαυμάσια. Ιδίω ε, όσον, όσον αφορά την καθημερινή επιβίωση νομίζω ότι ο ανταγωνισμός έχει δημιουργήσει μεγάλες τρευλώσεις και ότι υποφέρουν, υποφέρει η ύπεθρος και η επαρχία από αυτές τις τρευλώσεις. Ιδίω πιστεύω ότι η, όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές συνθήκες θα πρέπει να είναι κανείς πιο προσεκτικός. Θα πρέπει η φροντίδα, η φροντίδα το, για τους πολίτες, οι υπηρεσίες ε, φροντίδας και υγείας να λειτουργήσουν καλύτερα. Εκεί δεν νομίζω ότι ο ανταγωνισμός έχει επιφέρει σωστά αποτελέσματα. Επίσης υπάρχουν άλλες απόψεις ε, που λένε ότι και η συνεργασία μπορεί να δώσει το έναυσμα μιας ε, βελτίωσης ε, της ζωής και ότι η συνεργασία δεν πρέπει να υπόκειται στις επιταγές του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός έχει θετικές πτυχές αλλά έχει, μπορεί να επιφέρει και πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Λοιπόν πρέπει να υπάρχει απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ανταγωνισμού και συνεργασίας η οποία πρέπει να είναι δεδομένη και να εδρεωθεί. Εμείς προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις για τον ανταγωνισμό με τις τροπολογίες μας. Τώρα, για τις χρηματοοικονομικές αγορές σε αυτό το τμήμα ε, προσπαθήσαμε λίγο να τονίσουμε την έκθεση Βικάνεν και τα σημεία τα οποία ταιριάζουν με τις δικές μας απόψεις και παραπάνω Πέμπουμε επίσης και σε άλλους τομείς που πρέπει να συμπεριληφθούν στο θέμα του ανταγωνισμού. Ο τρίτος βασικός τομέας είναι τα τρόφιμα και η αγροτική πολιτική και γι' αυτό υποβάλαμε μία τραπολογία διότι πιστεύουμε ότι είναι κρίμα ότι όλη, όλη αυτή η κερδοσκοπία που γίνεται με τα τρόφιμα δεν έχει δελεχώς εξεταστεί και συμπεριληφθεί στην έκθεση. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτή την κερδοσκοπία που γίνεται στα τρόφιμα. Επίσης ε, τονίζουμε ότι στην Ομοσπονδιακή Γερμανία υπάρχουν μειώσεις τιμών, ναι, έχουν γίνει, αλλά έχουμε και αρνητικά ε, αποτελέσματα, αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι γίνεται μια μείωση τιμών, αλλά αυτή συμβαίνει εις βάρος της ποιότητας, υποφέρει ποιότητα των προϊόντων εν συνεχεία. Άρα λοιπόν και εδώ πάλι επιβάλλεται μια ισορροπία, η οποία δεν πιστεύω να εκφράζεται παρκώς στην, στην έκθεση και ε, στην, στον αγροτικό τομέα και στον προσανατολισμό της αγοράς του αγροτικού τομέα και εκεί δεν είμαι βέβαιος ότι ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι η μία και μόνη αρχή το ένα και μόνο κριτήριο. Υπήρχαν εποχές στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη πριν από αρκετούς αιώνες όταν ε, επλήγει ο πληθυσμό ε, μαζικά ε, λόγω έλλειψης τροφίμων ή καταστροφής ας πούμε κάποιου βασικού βασικής καλλιέργειας. Ε, έχουμε τέτοια παραδείγματα και δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στις δυνάμεις της αγοράς. Πρέπει να δούμε και έξω από αυτό το στοιχείο ε, έτσι ώστε κάθε παραγωγή να προσανατολίζεται στις αγορές. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή έχει υπερβολικά τονίσει όλες τις πτυχές του ανταγωνισμού και όχι τόσο τη συνεργασία και όλες τις άλλες πτυχές που ε, και αυτές συνάδουν στη βελτίωση του ανταγωνισμού. Η πρόεδρος, η Εύα. Ο, α, όχι. Ποιος? Είναι 6 παρα 10 και βλέπω να είναι αραιές οι τάξεις των βουλευτών. Θα περιοριστώ σε κάποια σχόλια μονάχα. Δύο σημεία τα οποία για μένα είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Και το θέμα αυτό σας λέω είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα γιατί βρισκόμαστε μέσα σε μια μεγάλη κρίση και είναι η στιγμή στην οποία συζητούμε για επίπεδα ανεργίας τα οποία είναι πια τρομακτικά. Η πρώτη παρατήρησή μου έχει να κάνει με την ε, έννοια του ανταγωνισμού, το αν είναι υγιής ή όχι ο ανταγωνισμός. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν υπόκειται σε υπερβολική γραφειοκρατία, κάτι που ανέφερε ο Ντέρκ και ο Γκίναρ. Θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποια σχόλια, λοιπόν, κατά την άποψή μου, για το περιορισμό της γραφειοκρατίας, τον απαραίτητο περιορισμό της γραφειοκρατίας και που θα μπορέσει να οδηγήσει σε καλύτερο ανταγωνισμό, σε περισσότερο ανταγωνισμό. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι κάτι που ανέφερε ο Γκούναρ. Οι κρατικές επιδοτήσεις μπορούν να καταστρέψουν τον ανταγωνισμό, το κατανοώ αυτό που αναφέρεις, αλλά συγχρόνως οι κρατικές επιδοτήσεις έχουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα στον υγιή ανταγωνισμό. Και πιστεύω γενικά ότι ο ανταγωνισμός οδηγεί εν καιρό σε χαμηλότερη ανεργία. Αυτά είναι τα δύο σημεία τα οποία θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα και θα ήταν χρήσιμο πιστεύω να βρίσκονται στην έκθεση του κ. Πεσέδο. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Νομίζω ότι όλοι έχουν μιλήσει. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Αντολίν. Ναι, ναι. Ο Σάλβα δεν θέλω να λάβει το λόγο. Ναι, πράγματι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο, κυρίως αυτοί που κατέθεσαν τροπολογίες και οι συνάδελφοι που έχουν συμμετάσχει στη σημερινή συζήτηση. Θέλω να επικροτήσω το επικοδομητικό τους πνεύμα και τις συμβολές τους, οι οποίες αξίζουν να ληφθούν υπόψη. Ε, για τις 120 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είχαμε καταρχήν 51 σημεία στα οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν συζητήσεις. Για μερικά από αυτά έχουμε τροπολογίες και έχουν προσθεθεί και ορισμένε νέες παράγραφοι. Ε, και φυσικά και ο κάθε έχει ένα περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων και λέξεων για να μπορέσει να, να αναφερθεί στην έκθεση της Κομισιόν. Να σταθώ στις παραγράφους που είχαν τις πιο πολλές τροπολογίες. Μία πρώτη τέτοια παράγραφος <clears throat> αφορά την κατάσταση της κρίσης που διατρέχουμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς για τις επιδοτήσεις που δίδονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα και συμμερίζομαι αυτά που είπε ο κύριος Έπινγκ ότι πρέπει να είναι περιορισμένε στον χρόνο αυτές οι επιδοτήσει και να έχουν ένα αναλογικό χαρακτήρα. Επίσης, για τις κρατικέ επιδοτήσει προ τράπεζες που απαιτούν, που χρειάζονται βοήθεια, υπάρχει μια πλειάδα τροπολογιών που θέλουν να απαλείψουν την αναφορά σε συγκεκριμένες τράπεζες. Από την άλλη μεριά είναι απαραίτητο να οι τράπεζες αυτές να προχωρήσουν σε σχέδια αναδιάρθρωσης που θα εξασφαλίσουν ότι θα ευδοκιμήσουν αυτές οι επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις αυτές δίνουν πλεονεκτήματα σε τράπεζες εάν δεν τις χρειάζονται πράγματι και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ισόπεδο γήπεδο ανταγωνισμού και ίση μεταχείριση για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα συμπεράσματα της ε, διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Επίσης, έχουν αναφερθεί ιδίως από τον κύριο Χιόκμαρκ τα θέματα των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητικός ο κύριος Χιόκμαρκ. Εδώ υπήρχαν αποκλίνουσες απόψεις σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι υπηρεσίες ε, γενικού οικονομικού συμφέροντος θεωρείται ότι πρέπει να εξαιρούνται από τους κανόνες του ανταγωνισμού Ορισμένοι θέλουν λοιπόν μια ευρία εξαίρεση, άλλοι θέλουν να έχουν μια πολύ περιορισμένη εξαίρεση. Το γεγονός όμως ότι υπάρχουν κρατικές επιδοτήσεις σε υπηρεσίες γενικού ε, οικονομικού συμφέροντος δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να τις εξαιρέσουμε συλλήδιν και να αυξήσουμε το κόστος ή να δημιουργήσουμε ε, ουσιαστικά αναποτελεσματικότητες στην παροχή αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια σωστή διαχείριση σε οικονομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και να βρούμε μια λύση. Επίσης υπήρξαν και κάποιες προτάσεις για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στα τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, για τις ε, φαρμακευτικές εταιρείες, για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά έχουν τύχει συνένεσης μεταξύ μας. Επίσης έχουμε το θέμα των συλλογικών ε, αγωγών όπου έχουν κατατεθεί και εκεί τροπολογίες. Νομίζω ότι αυτό μας έχει απασχολήσει εδώ και κάποιο διάστημα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να παρουσιαστούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα θέματα των συλλογικών αγωγών, να καταλήξουμε σε κάποιο είδου συμφωνία, ώστε το ζήτημα αυτό να πάρει σάρκα και οστά. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό που ανέφερε ο κύριος Χέκμαρκ είναι ο ρόλος της, του ανταγωνισμού στην πραγματική οικονομία. Ο κύριος Έπινγκ επίσης αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ο κύριος Κλούτε επίσης. Για μένα είναι σαφές ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να ευνοήσει μια πιο ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων και προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως στην έκθεση αυτή είναι να υπογραμμίσουμε το ρόλο που επέχει η πολιτική ανταγωνισμού για να αυξήσει και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να συμβάλλει στη στρατηγική 2020 για την ε, <clears throat> βιώσιμη ανάπτυξη και επίσης να υπάρξει η σωστή αντιμετώπιση των κρατικών κανόνων για να διατηρήσουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε υγιή κατάσταση σε μια στιγμή που υπάρχει τεράστια πίεση πάνω τους. Να έχουμε λοιπόν μια μεγαλύτερη προσοχή και αυστηρότητα σε σχέση με τις πολιτικές της, ε, των δημοσίων επιδοτήσεων γιατί τελικά είναι ο απλός πολίτης ο φορολογούμενος από την τσέπη του οποίου βγαίνουν τα χρήματα τα οποία θα πάνε σε αυτές τις επιχειρήσεις εγώ θέλω να πω ότι συμμερίζομαι αυτές τις ανησυχίες, υποστηρίζω τις προτάσεις αυτές και θα προσπαθήσω να βρω κάποια διατύπωση η οποία θα οδηγήσει σε συμφωνία μεταξύ όλων μας. Σε σχέση με το θέμα της κοινή αγροτικής πολιτικής, κύριε Κλούτε, εσείς είπατε ότι η ΚΑΠ δεν μπορεί να έχει μονάχα σαν στόχο την ε, ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων και των αγροτικών επιχειρήσεων. Στην έκθεση αυτή εγώ προσπάθησα να κάνω σαφής ότι ναι, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα η αγροτική πολιτική, αλλά πολλές φορές υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά αγροτικών προϊόντων και είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πολιτική σωστή σε ανταγωνιστικό επίπεδο, να υπάρξει όση ανταγωνιστικότητα μπορεί να υπάρχει στην, στην αγροτική πολιτική, γιατί αυτό θα είναι και προς το συμφέρον των καταναλωτών και προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, χωρίς να τεθεί ένα αμφιβόλο το πλέγμα των άλλων στόχων της κοινή αγροτικής πολιτικής, θα πρέπει πιστεύω να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τρόπους για να έχουμε ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Επίσης οι τροπολογίες που αφορούν το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρο... Ε, Κεντρικής Τράπεζας και οι νομισματικές πολιτικές των Τις τράπεζες αυτής έχουν σαν στόχο να διατηρήσουν τις ε, αγορές σε μια κατάσταση η οποία θα είναι προς το συμφέρον όλων των ε, ε, επιχειρήσεων. Είναι χρήσιμο λοιπόν να υπογραμμίσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων συστημικών φορέων που είναι πάρα πολύ σημαντικοί ώστε να τις αφήσουμε να καταρρεύσουμε. Επομένως χρειάζεται κάποια έμεση εγγύηση για τις επιχειρήσεις αυτές και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την επιβίωσή τους μέσα σε ισορροπημένες συνθήκες ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα θέματα ούτως ή άλλως θα τα αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της έκθεσης Λίκανεν. Ίσως θα μπορούσαμε εδώ να έχουμε και κάποια μνήα της έκθεσης αυτής, η συζήτηση για την οποία ήδη μόλις ξεκινάει τώρα για τις κρατικές επιδοτήσεις επίσης σας είπα ότι υπάρχει και μια ομάδα εργασίας που αντιμετωπίζει αυτές τις τροπολογίες και ο στόχος μας ήταν να έχουμε και ένα ψήφισμα για την απαραίτητη διαδικασία εξυγχρονισμού που λαμβάνει χώρα εφέτος. Όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις λοιπόν που αφορούν το πλαίσιο για τις κρατικές ε, επιδοτήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας να καταλήξουμε και σε μια συνολική θέση, ένα ψήφισμα το οποίο να εκφράζει τις απόψεις του Κοινοβουλίου για τον τομέα των κρατικών επιδοτήσεων και εν κατακλείδα, εν κατακλείδη, υπάρχουν ε, όλες αυτές οι τροπολογίες που νομίζω στην μεγαλύτερη πλειοψηφία τους μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο συμβιβαστικών λύσεων στο βαθμό του δυνατού και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινού για να καταλήξουμε σε μια έκθεση περί ανταγωνισμού η οποία να είναι ισορροπημένη και η οποία να τονίζει ιδιαίτερα το ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού στη γενικότερη οικονομική ε, δραστηριότητα και θα μπορέσει να συμβάλλει σε μια ευφυά και βιώσιμη αλλά και περιεκτική μορφή ανάπτυξη. Και επομένω, μέσα στα πλαίσια αυτή τη προοπτική, έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο η πολιτική ανταγωνισμού. Uh, σε ευχαριστούμε πολύ, Αντολίνο Αγκούνε. Νομίζω ότι θέλει να επανέλθει σε ένα σημείο. Παρακαλώ. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μακρηγορήσω, αλλά καθότι κάνουμε μια πολύ ευχάριστη συζήτηση αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να πω κάποιες ιδέες για τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες αναφέρθηκε στη δυνατότητα που αναφέρθηκε ο Συγητή, Όταν μιλάμε για υπηρεσίες οικονομικού, γενικού οικονομικού συμφέροντος, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι πολίτες αυτοί, οι οποίοι εξαρτώνται περισσότερο από αυτές τις υπηρεσίες, είναι οι πολίτες, οι, οι πολίτες αυτοί που θα πρέπει να έχουν και τι καλύτερε δυνατέ ευκαιρίε, ακριβώ επειδή εξαρτώνται από αυτέ τι υπηρεσίε. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να εξαιρούνται οι άνθρωποι αυτοί από τη δυνατότητα να επιλέξουν, να επιλέξουν ουσιαστικά την υπηρεσία με την καλύτερη ποιότητα. Και όπως ακριβώς είπε και ο συγητή, αυτό αποτελεί ένα απόσπατο στοιχείο του ισότιμου επίπεδου ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες θα πρέπει τελικά να επιδοτούνται και να βοηθούνται. Στόχος μας θα πρέπει να είναι περισσότερο οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πολίτες δηλαδή αυτοί να ενισχυθούν μέσω της νομοθεσίας αυτής, προκειμένου να έχουν την πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά και ένας πιο υγιής ανταγωνισμός και μια μεγαλύτερη γκάμα διαφορετικών υπηρεσιών, αν θέλετε, μεγαλύτερη επιλογή για τον ίδιο τον πολίτη. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουμε ήδη δει ότι ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι τάσσονται πλέον κατά τον ανταγωνισμό. Να θυμάστε, πριν από αρκετά χρόνια υπήρχαν πάρα πολλοί εκπρόσωποι πολλών πολιτικών ομάδων που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την τα μονοπόλια τα οποία υπήρχαν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, θεωρώντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα κατάφεραν να εξασφαλίσουν τι καλύτερε δυνατέ υπηρεσίε. Νομίζω, όπως είπε και ο εισηγητής, ότι θα καταφέρουμε, αν εντάξουμε και τις ιδέες αυτές, να έχουμε ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά και ποιοτική παροχή υπηρεσιών για όλους τους πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο για τη διευκρίνηση αυτή που ανέφερε για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες ουσιαστικά εξυπηρετούν την έννοια του, του πολίτη σε ένα κράτος. Δεν είναι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τις αγορές, αλλά είναι υπηρεσίες που αποτελούν τμήμα της ευθύνης ενός κράτους προς τους πολίτες του. Δεν θέλουμε όμως αυτές οι υπηρεσίες να έχουν υπερβολική τιμολόγηση ή να έχουν υπερβολικά έσοδα και κέρδη. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει δημόσια υποστήριξη, αλλά υπάρχουν στοιχεία τα οποία εμεί δεν μπορούμε να επηρεάσουμε γιατί εμπίπτουν στην πολιτική τη επικουρικότητα, στην επικουρικότητα των κρατών μελών. Απλώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει αναζήτηση τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα από την πλευρά των επιχειρήσεων και να δώσουμε μια δυνατότητα να υπάρχει καλύτερη επιλογή και ανταγωνιστικότητα αυτών των υπηρεσιών μεταξύ τους. Επομένως νομίζω ότι αυτό το οποίο αναφέρει και ο κύριος Χέρκμαρκ είναι μια σωστή και ισορροπημένη πρόταση. Εγώ θα προσπαθήσω να έχω μια συμβαστική πρόταση η οποία να λαμβάνει υπόψη αυτά τα οποία απασχολούν τον κύριο Χέρκμαρκ και ελπίζω θα γίνει και αποδεκτή και από τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Δεν έχουμε ακόμα χρονοδιάγραμμα για την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. <clears throat> θα μπορούσε να γίνει ψηφοφορία αυτή τον Ιανουάριο. Αυτά εξαρτώνται από το τι θα κάνουμε, τι θα αποφασίσουμε να κάνουμε με την έκθεση πρωτοβουλίας και την ε, χρονική της αλληλουχία. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι συντονιστές, γιατί πρέπει να απεληθεί στον επιτρεπόμενο αριθμό εκθέσεων πρωτοβουλίας. Όπως πάντα, εγώ προσπαθώ να προτείνω προς την συνέλευση των πρόεδρων των πολιτικών ομάδων ότι οι αιτήσει εκθέσει μα θα πρέπει να εξαιρούνται από τον αριθμό των ε, εκθέσεων πρωτοβουλία ώστε να μην περιορίζουν τον αριθμό που ε, μπορούμε να κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά προς το παρόν δεν το έχουμε πετύχει ακόμα και γι' αυτό θα περιμένουμε για τις συμβαστικές προτάσεις του Αντολίν και θα δούμε στη συνέχεια ποιο είναι το καταλληλότερο χρονοδιάγραμμα για την συνέχεια της έκθεσης αυτής. Αυτά λοιπόν για σήμερα μπορούμε να το ονομάσουμε μια μέρα. Κλείνω τη συνεδρίαση.